η παρέμβαση των Εθνικών Κοινοβουλίων στο νέο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ρόλο νομοθέτησης τη στιγμή που υπάρχει συναπόφαση δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Υπάρχουν ορισμένες αιτιολογικές σκέψεις που είναι λυσιτελείς, διότι ε, άπτονται της νομοθετικής διαδικασίας και γι' αυτό θα πρέπει να εξεύρουμε μία εξισορρόπηση μέσα στο πνεύμα της συνθήκης ε, της Λισαβόνας, διότι θα πρέπει να υπάρχει και να ενδυναμωθεί και το νομοθετικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως και τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να παρέμβουν και γι' αυτό το δικαστήριο ορίζει το όλο ζήτημα μέσα σε, στα πλαίσια ε, των, των επιμέρους οριοθετήσεων και εμείς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις ε, νομικές, νομικής υφής σκέψεις. Τώρα, μετά από ορισμένε παρεμβάσεις, θεωρώ ότι η Ευρώπη τα τελευταία 10 ή 12 χρόνια έκανε αποφασιστικά βήματα ε, υπέρ αυτού του εγχειρήματος. Φτάσαμε στην ΟΝΕ, στην διεύρυνση και για όλα αυτά τα μεγάλα στοιχεία χρειαζόταν ένα νομικό αρχιτεκτόνημα για να φτάσουμε σε αυτή τη νέα Ευρώπη στην Ευρώπη της ΩΝΕ, τη διευρυμένη Ευρώπη και ούτω καθεξής. Περάσαμε και υπερβήκαμε σωρία ζητημάτων. Αυτό είπε και ο προλαλής σας, ο οποίος είπε ότι πολλές χώρες δεν θέλουν δημοψήφισμα. Αλλά ας θεωρήσουμε ότι αυτό το αρχιτεκτονικό οικοδόμημα πέρασε από πολλά προσκόμματα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και στις 2 ε, Οκτωβρίου έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα βασικό δημοψήφισμα. Εγώ σας μιλώ όμως υπέρ ε, μιας πλειοψηφίας η οποία θέλει να εφαρμόσει την συνθήκη της Λισαβόνας, όπου θέλουμε να λήξει αυτό αυτή η διαδικαστική κολυσιεργία που ίσχυε τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε ένα ενισχυμένο κοινοβούλιο με δημοκρατικές αρχές. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να διεκδικήσουμε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί αυτή η απόφαση κατά της Ευρώπης, διότι η απόφαση ορίζει το γεγονός ότι ο θεμελιώδης νόμος της ε, Γερμανίας είναι συμβατός με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό θα πρέπει να το διεκδικήσουμε αυτό. Αυτή η απόφαση δεν αμφισβητεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική ερμηνεία, διότι ακριβώς αυτό διεκδικούμε για να οικοδομήσουμε όλα ένα και περισσότερη Ευρώπη. Ευχαριστώ που μας ε, υπενθυμίσατε μία νομική αρχή που θεωρούσαμε ως δεδομένη. Αλλά ξεχάσαμε δηλαδή ότι η αιτιολογική σκέψη, οι αιτιολογικές σκέψεις της απόφασης δεν έχουν νομική ισχύ. Μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ε, συζήτηση στο όλο ερμηνευτικό εγχείρημα. Σέφλιν. Ε, Thank you, Chairman. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν αυτή η συζήτηση. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Έφυγε και ο κύριο Σέβεριν, αλλά είμαι ευγνώμων γιατί μας έδωσε αυτή την μεταμοντέρνα ιδέα για τους προοδευτικούς αναχρονιστές. Υπάρχει αρνητική πλευρά και ρίχνω πολύ εκεί την έμφαση και εγώ εκεί θέλω να την αποδώσω. Βέβαια δέχομαι ότι υπάρχουν και θετικά σημεία. Ξέρετε, υπάρχει ένα σημείο όπου η πολιτική και ο νόμος συναντιούνται και δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα. Η απόφαση της Καζούρη, και εγώ το κοιτάζω το θέμα από πολιτική σκόπια, φαίνεται να έχει ξεχάσει ότι δεν είναι νησί η Γερμανία, ότι συνδέεται στην υπηρετική Ευρώπη και ότι αυτή η απόφαση επηρεάζει, εν πάση περιπτώσει, ολόκληρη τη γυραιά Ήπειρο. Δεύτερον, πρέπει να προσθέσουμε το... την ερώτηση πού πρέπει να βασίζεται αυτό το Σύνταγμα και πώς πρέπει να κατοχυρώνουμε την εκπροσώπηση μέσα σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω από την απόφαση και ευχαριστώ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 et puis les compétences européennes, qu'il s'agisse de compétences communautaires, voire même fédérales, s'agissant de la monnaie, communautaires pour beaucoup de politiques. Et, Όταν πρόκειται για το ενιαίο νόμισμα. Διότι έχουμε να κάνουμε και με διακυβερνητικές αρμοδιότητες ή απλή συνεργασία. Νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα διατρέχουμε το κίνδυνο αυτής της ε, σύγκρουσης και όπως είπε και ο Γκίφερ Χόφστατ και ο Μέντες Δεβίγκο, πέρα από τις συζητήσεις που έχουμε σήμερα και ξέρουμε ότι σε άλλες χώρες, άλλα συνταγματικά δικαστήρια μπορούν να γνωμοδοτήσουν ή να λάβουν αποφάσεις, και θα πρέπει να φτάσουμε στα σωστά ε, συμπεράσματα. Μιλάμε για την δημοκρατική διαδικασία, για την συνομιλία με τους πολίτες και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι η ΑΦΚΟ θα έπρεπε να προτρέχει των γεγονότων του τι μπορεί να συμβεί στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες και θα μπορούσαμε να προκαλέσουμε στην πενταετία αυτή σε κάθε πρωτεύουσα να προκαλέσουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό της ε, συγκατοίκησης ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων με εθνικές. Κάποια στιγμή που οι πολίτες θέτουν πολλά ερωτήματα, όπως είδαμε στις ευρωεκλογές. Με βάση λοιπόν αυτή την προειδοποίηση της γερμανικής απόφασης θα πρέπει να προτρέξουμε και να άρουμε αυτές τις ε, ε αναρμοδιότητες ή την έλλειψη κατανόησης ενός κειμένου. Εμείς θέλουμε να εγγράψουμε αυτές τις έννοιες στη νέα συνταγματική μας συνθήκη. Θα θέλαμε λοιπόν η δική μας Επιτροπή να προτείνει σε κάθε πρωτεύουσα για την επόμενη πενταετία σε επίπεδο αρμοδίων, σε επίπεδο νομομαθών, σε επίπεδο ε, κοινωνίας των πολιτών ή εθνικών κοινοβουλίων, να προτείνουμε δημόσιες συζητήσεις για να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα, γιατί δεν φοβόμαστε αυτά τα ερωτήματα έναντι μίας γενικότερης δημοκρατίας και δημοκρατικών θεσμών. Φτάνουμε στα συμπεράσματά μας. Η κυρία Γιαννάκου. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάναμε σήμερα ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες χώρες ή σε σχεδόν όλες το ευρωπαϊκό δίκαιο θεωρείται ότι υπερέχει του εθνικού. Εμείς στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη, δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο. Υπάρχει όμως ανώτατο δικαστήριο που έχει δικαίωμα να κρίνει τη συνταγματικότητα των νόμων και ούτω καθεξής. Μέχρι σήμερα δεν έχει αγγίξει το θέμα αυτό στα ζητήματα που αφορούν στις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων ε, με την προσπάθεια ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Εάν η απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου αποτελέσει προηγούμενο για όλα τα συνταγματικά ή ανώτατα δικαστήρια που υπάρχουν στις ε, διάφορες χώρες, τότε η υπόθεση αυτή φεύγει από το πολιτικό της περιεχόμενο. Παραδείγματο χάρη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαστηρίου σε ποιο βαθμό αντιλαμβάνεται τη συνεργασία που μπορεί να κάνει το γερμανικό κράτος ή στις πολιτικές αποφάσεις που μπορεί να λάβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε συνεργασίες με τρίτες χώρες. Διότι εδώ δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά δική της νομική οντότητα. Βεβαίως αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο έχει μια ιστορία. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε ως ανάχωμα σε πιθανές εξελίξεις μετά τον πόλεμο που θα παρομοίαζαν με αυτές του Τρίτου Ράιχ ήταν ο λόγος για τον οποίο έγινε το συνταγματικό δικαστήριο. Δηλαδή είναι τελείως άλλοι λόγοι για τους οποίους έγιναν ανώτατα οι συνταγματικά δικαστήρια σε άλλες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να μεταθέσουμε μια αμυγός πολιτική υπόθεση και να την αφήσουμε σε χέρια νομικών και συνταγματολόγων. Είναι σωστό βεβαίως οι νομικοί μας σύμβουλοι να κάνουν την ανάλυση του ζητήματος αλλά έχω την εντύπωση ότι αντί να φροντίσουμε να διαχυθεί αυτό σε όλη την Ευρώπη, καλό θα ήταν να το περιορίσουμε στα γερμανικά όρια, διότι η γερμανική κυβέρνηση και οι γερμανικές πολιτικές δυνάμεις είναι υπεύθυνε για το πώς και θα προσαρμοστούν στις πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν και που είναι η συνθήκη της Λισαβόνας και άρα ο πρόεδρός τους θα καταθέσει το αντίστοιχο έγγραφο και θα δημιουργήσουν ένα θεμελιώδη συνταγματικό νόμο ο οποίος θα είναι ανάλογος. Άλλωστε και τα συντάγματα αλλάζουν. Δηλαδή, αν μιλάμε για το μέλλον, αν μιλάμε για αυτά που θέλουμε να κάνουμε, τα συντάγματα δεν μένουν ίδια. Εμείς αλλάξαμε το σύνταγμα, η Ιταλία έχει αλλάξει το σύνταγμά της πρόσφατα και πάρα πολλές άλλες χώρες. Τίποτα δεν μένει αμετακίνητο. Νομίζω λοιπόν ότι με όλο το σεβασμό δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα σε αυτή την υπόθεση από όσοι της αξίζει. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Μπρόντς. Το Συνταγματικό Δικαστήριο παρά την ρητορική περί προστασίας της ε, εθνικής ε, κυριαρχίας κατ' ουσίαν υποστηρίζει τους ε, πολιτικούς με το εγχείρημα του αυτό αυταπατάται και θεωρεί πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται μια ομοσπονδιακή ένωση, ενώ αυτό ακριβώς κάνει. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί λέει πως μια τέτοια εξέλιξη απαιτεί μεγάλες συνταγματικές αλλαγές και ακόμα και δημοψήφισμα, κάτι το οποίο βεβαίως οι πολιτικοί δεν θέλουν και είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει συμβεί και στις 27 χώρες. Το συνταγματικό δικαστήριο παριστάνει ότι επικρίνει την διάβρωση των εθνικών εξουσιών, αλλά με το να λέει πως, αλλά με το να πως συνθήκη τη Λισαβόνα δεν είναι αντίθετη με το Γερμανικό Σύνταγμα, δίνει το πράσινο φω στη συνθήκη τη Λισαβόνα και άρα στην Ομοσπονδιακή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Ε, Τελευταία παρέμβαση. Όχι, όχι, όχι, όχι. Τελειώσαμε με τους ομιλητές, λέει ο πρόεδρος. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον νομικό σύμβουλο ή από τον συνεργάτη του να μας απαντήσουν σε αυτές τις υποδείξεις όπως ανέκυψαν από την παρούσα συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως η συζήτηση κατέδειξε πόσο σημαντικό είναι να γίνει συζήτηση για τη σχέση του Εθνικού Συνταγματικού Δικαίου με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η τελευταία μεγάλη συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε χώρα πριν από 16 χρόνια ε, με αφορμή την απόφαση του Γερμανικού Σταγματικού Δικαστηρίου για τη συνθήκη του Μάστριχτ. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια παρακάτω, περαιτέρω φάση της ευρωπαϊκής ε, ενοποίησης και έχουμε μια νέα απόφαση του Σταγματικού Δικαστηρίου όσον αφορά τη μελλοντική εξέλιξη της ενοποίηση. Σύντομα θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις για τα δύο βασικά σημεία αυτής της απόφασης. Πρώτα απ' όλα για το δημοκρατικό έλλειμμα. Θεωρώ πως το Συνταγματικό Δικαστήριο βλέπει εδώ πέρα μια εγγενή, εγγενή στο, ένα εγγενές στο σύστημα κενό το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό όμως γίνεται εφαρμόζοντας κριτήρια ενός κράτους σε ένα σύστημα το οποίο δεν είναι κράτος, είναι ένας ιδιόμορφος διεθνής οργανισμός. Και έχουμε βεβαίως το εθνικό και το ε, διεθνές δίκαιο και όχι κάποιο, ίδιο, κάποιο τρίτο είδος βεβαίως θα μπορέσουμε να έχουμε μια, μια διαφορετική κατανομή, θα μπορέσουμε να προσφέρει και μια διαφορετική λύση. Έχουμε ένα μεικτό σύστημα, ένα κοινοβούλιο και ταυτόχρονα εκπροσώπηση των κρατών, το οποίο όμως έχει εξίσου ισχυρή δημοκρατική νομοποίηση όπως ε, ένα οποιουσδήποτε άλλος, οποιαδήποτε άλλη κρατική οργάνωση. Και βεβαίως ε, ακούσαμε και την ερμηνεία του κυρίου Φερχόφστατ πως η λύση θα μπορούσε να είναι μια ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως το δικαστήριο το βλέπει αλλιώς. Εδώ πέρα μιλάει για ενίσχυση της συναπόφασης των εθνικών κοινοβουλίων στην διαδικασία αυτή. Τώρα αν αποτελεί λύση αυτό δεν ξέρω. Δεύτερο στοιχείο της συζήτησης ήταν τα δικαιώματα του Συνταγματικού Δικαστηρίου να ασκεί έλεγχο. Το πώς, το πού θα φτάσουν θα το δούμε στο μέλλον. Στην πράξη δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ε, προβλέψεις ε, τι θα γίνει εάν θα έχει τον τελικό λόγο το Συνταγματικό Δικαστήριο θα ε, συμβεί αυτό κάτι τέτοιο μόνο αν έχουμε ακραίες περιπτώσεις ή όπως λέει και το ίδιο το δικαστήριο εάν συμβεί κάτι και αλλάξει η δικονομία του ιδίου, του ιδίου δικαστηρίου για να μπορέσει να ασκήσει αυτόν τον έλεγχο τον οποίο επιζητεί. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει ο κίνδυνος το μέσο αυτό να χρησιμοποιείται περισσότερο στο μέλλον, δηλαδή να έχουμε υποθέσεις οι οποίες θα φτάνουν ενώπιον του δικαστηρίου περί ε, υπέρβαση των αρμοδιοτήτων των ευρωπαϊκών οργάνων. Πράγματι, ο κύριος Μέσερ Σμιτ ε, ε, έχει δίκιο. Όταν αποφασίσει ένα δικαστήριο, όταν μιλήσει ένα δικαστήριο, μίλησε η Καλσρούη, η υπόθεση τελείωσε. Αλλά βεβαίως και το δικαστήριο δεσμεύεται από τις δικές του τις αρμοδιότητες γιατί υπάρχει το ευρωπαϊκό δίκαιο το οποίο ορίζει τις αρμοδιότητες και είναι πράγματα τα οποία έχει εγκρίνει το ίδιο το συνταγματικό δικαστήριο. Το εάν δηλαδή θα αναλάβει κάποιες αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο θα κρίνει αποκλειστικά το ΔΕΚ. Και ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η μελλοντική σύγκρουση είναι το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο να τηρήσει την υποχρέωσή του την οποία ε, το ίδιο ενέκρινε στην απόφαση περί Μάστριχτ περί συνεργασίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα αίτημα της Καλσρούης προς το Λουξεμβούργο. Άλλα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια το έχουν κάνει και έχει υπάρξει μια σχέση συνεργασίας και το House of Lords, της, το Βρετανικό Ανώτο Δικαστήριο. Μέχρι στιγμής από την Καλσρούη δεν υπάρχει τέτοια διάθεση. και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει για να μην υπάρξει τέτοια σύγκρουση στο μέλλον. Επίσης, ε, να σας πω πως η νομική υπηρεσία ήδη προετοιμάζει την ε, γνωμοδότησή της, ε, έχει υποβληθεί στην Σύνοδο των Προέδρων ήδη και θα είναι και στην διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ε, κλείνει η συζήτηση απόψε, αλλά νομίζω ότι φτάνουμε σε ορισμένα συμπεράσματα καταρχήν. Οι αιτιολογικές σκέψεις δεν μας δεσμεύουν από νομικής πλευράς. Οι αιτιολογικές σκέψεις μας δίνουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε αυτή τη θεματική. Άρα θα δράξουμε την ευκαιρία για να συζητήσουμε τα ζητήματα που ανακύπτουν. Κανένας δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα της Γερμανίας, ούτε να αλλάξει την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Πρόκειται για μια πολιτισμική διαδικασία εμβάθυνσης, την οποία μπορούμε να προβούμε και να λάβουμε υπόψη αυτή, αυτές τις επιμέρους πραγματικότητες των λαών. Και πέρα από τη γραπτή έκθεση, που ζητήθηκε από την νομική υπηρεσία, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε αυτή την ιδέα όπως ανέκυψε από τη συνάντηση των συντονιστών αλλά και από την ε, Επιτροπή μας να οργανώσουμε μια μεγάλη ακρόαση επί του θέματος αυτού. Τώρα με τους συντονιστές θα δούμε κατά πόσο μπορεί να ε, γίνει κάτι τέτοιο, να υλοποιηθεί. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς να καλέσουμε τους ε, δικαστές του συνταγματικού είτε από τη Γερμανία είτε από άλλα δικαστήρια. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να καλέσουμε συνταγματολόγους που είναι οι θύνοντες επί του θέματος και να μας πούνε πώς έχει το συνταγματικό ζήτημα στην εκάστοτε χώρα. Ας περάσουμε λοιπόν στο έκτο, μάλλον το πέμπτο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης που αφορά την προσαρμογή του κανονισμού στη συνθήκη της Λισαβόνας. Στις 21 Ιουλίου είχαμε αποφασίσει υπέρ των ε, προπαρασκευαστικών διαδικασιών και ορίσαμε ως συγητή τον David Μάρτιν. που αντικαθιστά τον κύριο Κόρμπετ. Είχε γίνει, μία, μάλλον ελήφθη μία πρώτη απόφαση στην προηγούμενη θητεία επί του θέματος, αλλά οι εργασίες έληξαν λόγω λήξης της θητείας, άρα ο συνάδελφος ε, Μάρτιν σήμερα θα μας παρουσιάσει την, ε, τις εργασίες αυτές και έλαβε υπόψη και τις εργασίες της Επιτροπής κατά την προγενέστερη θητεία. Έχει το λόγο ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για το ότι ο κύριος Σούν στην συζήτηση που προηγήθηκε ανέφερε την συνθήκη του Μάστριχτ και τις συζητήσεις που είχαμε με το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο γιατί επειδή είμαι εδώ πέρα πάνω από δεκαετία, νομίζω ότι βλέπω το ίδιο έργο ξανά και ξανά με τις αποφάσεις του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, αλλά χαίρομαι που ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μια καινούρια απόφαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ξανά στην Επιτροπή, αν και είναι λίγο γλυκόπικρη η κατάσταση, γιατί βρίσκομαι εδώ μόνο επειδή ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ, που ήταν εξαίρετο μέλος της Επιτροπής και ειδικό στα συνταγματικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς έχασε την έδρα του στις εκλογές. Όπως είπατε κάτω ουσίαν έχω την έκθεση του Ρίτσαρτ και έχω κάνει τρεις ε, αλλαγές. Να πω πριν περάσουμε ουσία πως πρέπει να καταστήσω σαφές, δεν ξέρω αν συζητήθηκε τον Ιούλιο, πως με την έκθεση αυτή δεν προδικάζουμε το τι θα γίνει, δεν κάνουμε καμία υπόθεση για το τι θα γίνει ε, με το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία. Απλά προετοιμαζόμαστε για κάποιο γεγονός που μάλλον είναι ε, προβλέψιμο και θα ήταν λάθος εκ μέρους να μην προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο να τεθεί της, ε, σε ενισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν λοιπόν, προδικάζουμε τίποτα, απλά είμαστε προετοιμασμένοι. Για να υπενθυμίσω λοιπόν στους παλαιούς συναδέλφους και, και για να μάθουν και οι Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ε, έκθεσης και τις τρεις ε, προσθήκες που ε, υιοθετήθηκαν 23 Απριλίου. Πρώτο νέο χαρακτηριστικό είναι ένα νέο άρθρο του κανονισμού για να μπορεί το Κοινοβούλιο να εξετάζει προτινόμενη νομοθεσία ε, για το εάν και κατά πόσον σέβεται τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχει αυτό συνθήκη Λισαβόνα, χρειάζεται και η ανάλογη διαδικασία. Δεύτερον, δεύτερη αλλαγή. Εισάγεται εδώ πέρα μία διαδικασία έτσι ώστε όταν ένα κράτος μέλος έχει αντίρρηση για κάποια νομοθετική πρόταση της Κομισιόν με βάση τις αρχές αναλογικότητας και της επικουρικότητας, ε, σύμφωνα βέβαια με τον νέο πρωτόκολλο για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, να μπορούμε να οργανωθούμε εντός Κοινοβουλίου, να υπάρξει κάποιος καταμερισμός εργασίας, δηλαδή το ζήτημα της ουσίας να πάει στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και το θέμα της ε, επικουρικότητας θα το κρίνει είτε η δική μας Επιτροπή είτε η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Και αυτές είναι οι λεγόμενες ε, κίτρινες και πορτοκαλί κάρτες έτσι έχει επικρατήσει να λέγονται, αλλά χρειάζεται μια διαδικασία και γι' αυτό. Και μετά έχουμε και ένα νέο κεφάλαιο που λέγεται συνταγματικά θέματα και έχουμε εδώ πέρα κάποια από τα νέα δικαιώματα που έχουμε αποκτήσει με την Συνθήκη της Λισαβόνας και κάποια που προϋπήρχαν π.χ. η πρωτοβουλία για την απλή και απλοποιημένη αναθεώρηση της συνθήκης που θα επιτρέπει σε ένα, πρωτοβουλία για να αποχωρήσει ένα κράτος μέλος από την Ένωση. Όλες αυτές είναι νέες διαδικασίες, όλα αυτά έχουν πάει σε ένα ενιαίο κεφάλαιο μαζί με υπάρχουσες συνταγματικές διατάξεις όπως ε, παραβίαση από κράτος μέλος ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αρχών τέταρτο χαρακτηριστικό της ε, συνθήκης που ευθύθηκε 22 Απριλίου είναι η προσαρμογή του κανονισμού όσον αφορά τον πρόεδρο της ε, Κομισιόν και βεβαίως ε, κυρίως την εκλογή αντί για τον διορισμό του και τον νέο τον είπα εκπρόσωπο, ο οποίος αλλάζει τίτλο και είναι είπα εκπρόσωπος για εξωτερικές υποθέσεις και πολιτική ασφάλειας και Λαμβάνεται υπόψη επίσης η δημιουργία νέου, ενός νέου νομοθετικού μέσου για να δούμε ποιος θα είναι ο έλεγχος που θα ασκήσει το Κοινοβούλιο για αυτό το α, παράγωγο δίκαιο. Όπως σας είπα όλα αυτά έχουν ήδη εγκριθεί από την προηγούμενη Επιτροπή Συνταγματικών Δικαιωμάτων. Εγώ έχω καταθέσει τρεις τροπολογίες ίσονος σημασίας για να ληφθεί υπόψη ότι έχει γίνει από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα. Πρώτα απ' όλα αφορά την απόφαση του δικαστηρίου που απαιτεί από εμάς να αιτιολογούμε τις αποφάσεις περί ασυλίας, άρσης ή μη, οπότε ε, αλλάζει ο κανονισμός για να ληφθεί αυτό υπόψη. Δεύτερη πρόταση για νέα τροπολογία, για να αλλάξουν τα άρθρα για τους παρατηρητές για να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Συμβουλίου της 18ης και 19 Ιουνίου οι συνάδελφοι που ήταν εδώ και στην προηγούμενη θητεία θα θυμούνται πως ε, είπαμε πως οι παρατηρητές είναι άτομα τα οποία θα είχαν εκλεγεί στο κράτος μέλος τους εάν ε, ε, ήταν, εάν γίνονταν ευρωεκλογέ και το κράτο μέλο. Αλλά το αλλάξαμε αυτό για να τσορίζει το κάθε κράτο μέλο με του δικού του κανόνε. Και τέλο, για να εκπροσωπείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή, την ΚΟΣΑΚ, την ε, Επιτροπή μεταξύ του Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και πως ο πρόεδρος δεν πρέπει να είναι πλέον αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής μας. Και πάλι είναι μια αλλαγή που... στην οποία συμφωνούν όλοι, υπάρχει γενική συνένεση και τα είχε προτείνει και ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Αυτό το οποίο μου προτάθηκε και εγώ δεν το υιοθέτησα, αλλά θα μπορούσαν ίσως να το δουν οι συντονιστές. Μου προτάθηκε το ζήτημα να δούμε το ζήτημα των αντιπροέδρων των επιτροπών. Ξέρετε πως κάθε επιτροπή έχει τέσσερις αντιπροέδρους Σύμφωνα με τον κανονισμό μας, εμείς θα έπρεπε να έχουμε μόνο τρεις. Το τροποποιήσαμε αυτό στην προηγούμενη θητεία, αλλά η τροποποίηση του κανονισμού ε, εξέπνευσε μαζί με την θητεία του προηγούμενου κοινοβουλίου και μου είπαν πως θα μπορούσα να αλλάξω τον κανονισμό. Υπάρχει πρόβλημα με την Συνδίκη της Λισαβόνας. Εάν θέλετε μπορεί να μπει και εδώ πέρα, ειδικά εάν το θέλουν και οι συντονιστέ, μπορεί να γίνει το εξή. Μπορούν να προτείνουν οι συντονιστέ να αλλάξει ο κανόνα από του τρει στου τέσσερι αντιπροέδρου. Η δική μου προτίμηση είναι να προτείνουν στην αρχή κάθε θητείας να προτείνουν ή να προτείνει η διάσκεψη των προέδρων, τον αριθμό των αντιπροέδρων της κάθε επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. E Ωραία. Ανοίγει η συζήτηση. Ο κύριος Ντάρφε. Ντάφ έχει το λόγο. Α, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, δεν είδα ένα όνομα. Μέντες Ο κύριος Μέντες Δεβίγκο ζήτησε το λόγο. Μία διασάφηση που δεν, κάτι που δεν κατανόησα. Εδώ στο έγγραφό μας, στα έγγραφά μας έχουμε το προσχέδιο του David Martin που φέρει ημερομηνία 28 Ιουλίου. Αυτό συζητάμε. Αυτές είναι οι τροπολογίες δηλαδή που εγκρίθηκαν από το προγενέστερο ε, κοινοβούλιο του Richard Corbett δηλαδή με, τα τρία, με τις δικές σας τρεις τροπολογίες. Άρα θα υπάρχει μια νέα προθεσμία υποβολή τροπολογιών από αυτή την Επιτροπή και θα ξαναψηφίσουμε ε, εδώ στην Επιτροπή και μετά θα πάμε στην Ολομέλη. Και το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει και τις δικές σας τρεις τροπολογίες. Ναι, ακριβώς. Θα πρέπει να ορίσουμε προθεσμία και θα ορίσουμε την ε, ημερομηνία ψηφοφορίας για να πάμε στην Ολομέλη. Ο κύριος Μέντες Δεβίγκο έχει δίκιο. Ένα επιπρόσθετο σημείο δεν θα υποβληθεί στην Ολομέλη αυτό το έγγραφο μέχρι ότου ξέρουμε ότι ενεκρίθη η συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά στα πλαίσια της Επιτροπής θα μπορούσαμε να ορίσουμε προθεσμία υποβολής τροπολογιών και στην Επιτροπή να εγκρίνουμε την έκθεση. Το ένα δεν αποτρέπει το άλλο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα και εγώ ε, να πω ότι είναι μεγάλη χαρά να... το γεγονός ότι ο Ντέιβιτ Μάρτιν ανέλαβε αυτή τη διαδικασία, πήρε τη σκητάλη δηλαδή. Είχε διατερματίσει σημαντικό ρόλο στη συνθήκη του Μάστρικτ και του Άμστερνταμ στις διασκέψεις εκείνες και αποτελεί κάτι παραπάνω από μία υποσημείωση στη διαδικασία αυτή της ε, οικοδόμησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανελικτικής της πορείας. Αλλά ε, Λυπάμαι διότι ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ δεν είναι παρόν, διότι ξέρουμε ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτω από ιδιάζουσες και δυσχερείς συνθήκες για να βελτιώσει τις πολιτικές συζητήσεις, τα πολιτικά ε, δρόμενα από ποιοτικής πλευράς. ως προς την, πολιτική τους, την ευρωπαϊκή τους διάσταση, αλλά φαντάζομαι ότι θα επανέλθει πριν ε, διανύσουμε ε, μακρύ χρονικό διάστημα. Άρα ας μην προβώ σε πολλές ε, ε, φιλοφρονήσεις, διότι όταν θα επανέλθει θα αρχίσουμε να μονομαχούμε, όπως κάναμε και στο παρελθόν. Τώρα, ως προς την έκθεση ενώπιών μας, βεβαίως θα μας απασχολήσει διεξοδικά μέσα από τις τροπολογίες αλλά υποθέτω ότι οι φιλελεύθεροι, οι άλτε, δεν θα υποβάλουν ουσιαστικές τροπολογίες. Είμαστε γενικά ικανοποιημένοι από την έκθεση αυτή στην ε, προγενέστερη της μορφή και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να είναι έτοιμο να είναι πανέτοιμο για να εφαρμόσει τη συνθήκη όταν θα παραστεί ανάγκη. Εάν αποτύχουμε στην σωστή προπαρασκευή, τότε εκτιθέμεθα σε επικρίσεις πολύ σωστά από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και από τους ίδιους τους πολίτες που εκπροσωπούμε. Μιλάμε για μια προπαρασκευαστική διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι προδικάζουμε την έκβαση του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία. Άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή αυτήν την έκθεση τη στιγμή που δεν μπορούμε να προδικάσουμε την έκβαση του δημοψηφίσματος. Αυτό ε, ήδη ελέγχθη ότι δηλαδή στην ε, υποβολή, η υποβολή μάλλον τροπολογιών βασίζεται στην προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η συνθήκη. Γενικά όμως δεν προδικάζουμε τα πράγματα. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε την ε, συζήτηση το αργότερο μέχρι τις 6 Οκτωβρίου. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να σας προτείνω την 16 Σεπτεμβρίου. 16 Σεπτεμβρίου στις 12 τη νύχτα. Τι λέτε, συμφωνείτε με αυτή την προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Ωραία. Θα συζητηθεί